Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε με τις ψηφοφορίες και θέτω σε ψηφοφορία την έκθεση του κυρίου Ρόντας για την κοινή αλλιευτική πολιτική. Πρώτα απ' όλα θέλω να θέσω σε ψηφοφορία 125 τροπολογίες της Επιτροπής Αλληλείας, όλες μαζί. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται τροπολογία αριθμός 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ θα ελέγξουμε Τροπολογία 4. Έλεγχος. Έναρξη του ελέγχου. Λήξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 5 έναρξη παρακαλώ λήξη εγκρίνεται τροπολογία 7 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν δεν σηκώνετε τα χέρια θα κάνουμε συνεχείς ελέγχους δυστυχώς. Τροπολογία 11. Έχετε δίκιο. Τροπολογία 7, το δεύτερο τμήμα υπέρ. Τροπολογία 7, το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε, να ελέγξουμε. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 7, έλεγχος. Λήξη. Εγκρίνεται. Ωραία, έχετε δίκιο. Να σηκώνετε τα χέρια σας για να μπορεί το Προεδρείο να βγάζει συμπεράσματα ασφαλή. Τροπολογία 11. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την τροπολογία 25. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Έλεγχος τροπολογία 48. Έναρξη του ελέγχου. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν μπορώ να βγάλω ασφαλέ συμπέρασμα. Έλεγχος 55. Έναρξη του ελέγχου. Λήξη. εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 60 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο τμήμα έλεγχος στο δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 60 έναρξη λήξη εγκρίνεται τρίτο τμήμα τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές έλεγχος τρίτο τμήμα της τροπολογίας 60 έναρξη λήξη εγκρίνεται τροπολογία 63 με ονομαστική κλίση έναρξη λήξη εγκρίνεται. Τροπολογία 72 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την τροπολογία 74. Έναρξη του ελέγχου. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος επί της τροπολογίας 81. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος επί της τροπολογίας 93. Έναρξη. Συνάδελφοι, να σηκώνετε τα χέρια σας. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται Τροπολογία 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 101 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παρακαλώ. Your micro, please. I'm sorry. I'm sorry for the house to take your... Λυπάμαι... With our internal... Λυπάμαι που σας απασχολώ για ένα εσωτερικό θέμα υπάρχει ένα, έγινε ένα σφάλμα. Στο πρώτο τμήμα του 106 ψηφίσαμε όχι και στο δεύτερο ναι. Συγγνώμη που, σας, ε, που πήρα το χρόνο. Έχουμε ψηφίσει την τροπολογία 101 σε δύο τμήματα. Θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία της τροπολογίας 106, έτσι κι αλλιώς. 106. Okay. We can repeat the vote. Δεν είχαμε ψηφίσει το 106. Το πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 107. Ε, Συγγνώμη, δεύτερο τμήμα τροπολογίας 106. Υπέρ. Υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε δεύτερο τμήμα της 106 έλεγχος έναρξη λήξη εγκρίνεται 107 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 116 υπέρ. Συγγνώμη, δεύτερο τμήμα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν χρειάζεται νομίζω αυτού του είδους ε, η συμπεριφορά. Δεν είμαστε σε γήπεδο κύριε συνάδελφοι. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 107 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 116 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 118 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται.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 αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ Θέλετε να ελέγξω την 142. Έλεγχος της 142. Έναρξη παρακαλώ. Λήξη. εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 179 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος επί του πρώτου τμήματος της 179 έναρξη λήξη εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έχω την εντύπωση περνάμε καταπίπτει το δεύτερο μέρος περνάμε στην τροπολογία 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 182 κατέπεσε εφόσον καταψηφίστηκε το πρώτο τμήμα τροπολογία 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα ελέγξουμε 195 έλεγχος έναρξη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 τέταρτο τμήμα της τροπολογίας 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 211 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 235 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται νομίζω να ελέγξουμε τη 235 παρακαλώ έναρξη. Λήξη. εγκρίνεται. τροπολογία 236 με ονομαστική κλίση έναρξη. λήξη. απορρίπτεται. Η τροπολογία 278 έχει αποσυρθεί και περνάμε στην τροπολογία 279. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 62 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 220 με ονομαστική κλίση έναρξη λήξη εγκρίνεται. Τροπολογία 280 Μονομαστική κλίση έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 237. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται να ελέγξουμε 237 έλεγχος λήξη του ελέγχου εγκρίνεται τροπολογία 246 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε. 246 έλεγχος. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 85 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος της τροπολογίας 85 έναρξη λήξη εγκρίνεται τροπολογία 247 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 248 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε τη 248 έναρξη λήξη απορρίπτεται τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 303 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 250 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 94 υπέρ κατά έλεγχος επί της τροπολογίας 94 έναρξη λήξη απορρίπτεται τροπολογία 290 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 221 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θέτω σε ψηφοφορία το αντίστοιχο τμήμα των τροπολογιών 215 και 281 με ονομαστική κλίση έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτονται. Τροπολογία 215 με ονομαστική κλίση, έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 281 με ονομαστική κλίση έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 251. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ελέγχουμε την τροπολογία 222 έναρξη λήξη απορρίπτεται τροπολογία 282 με ονομαστική κλίση έναρξη λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 291. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 304. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 252 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και περνάμε στην τροπολογία 282 με ονομαστική κλίση έναρξη λήξη απορρίπτεται Τροπολογία 283. Ονομαστική κλίση έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 284 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να ελέγξουμε τη 284 έναρξη του ελέγχου λήξη απορρίπτεται 253 με ονομαστική κλίση έναρξη λήξη απορρίπτεται τροπολογία 103 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θέτω σε ψηφοφορία το αντίστοιχο τμήμα της τροπολογίας 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 295 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε τη 295 έναρξη λήξη συγγνώμη έλεγχος της 295 έναρξη λίγη υπομονή Λήξη. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 295 καταπίπτει, συγγνώμη, η τροπολογία 104 καταπίπτει. Περνάμε στην τροπολογία 105. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 238 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ελέγχουμε τη 238 έναρξη λήξη απορρίπτεται 292 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 300 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 239 με ονομαστική κλίση έναρξη λήξη εγκρίνεται ψηφοφορία ε, τροπολογία 257 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 258 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 114 συγγνώμη τροπολογία 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 260 υπέρ κατά αποχές δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα έλεγχος στις 260 παρακαλώ έναρξη του ελέγχου λήξη εγκρίνεται τροπολογία 114 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος της 114 έναρξη λήξη εγκρίνεται τροπολογία 261 καταπίπτει τροπολογία 262 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 296 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 296. να ελέγξουμε τη 296 έναρξη του ελέγχου Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 297 με ονομαστική κλίση έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Ο εισηγητής έχει ζητήσει το λόγο για να προτείνει μια προφορική τροπολογία. Ο κύριος Ρόντους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εξ ονόματος της, ε, της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να υποβάλω την εξής προφορική τροπολογία ε, ε, στο άρθρο 15 παράγραφος 1 το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου του 2014 η αλία των μικρών πελαγικών ειδών, δηλαδή ε, σκουμπριά, ρέγγες, ε, σαρδέλες, σαφρίδια, παπαλίνες και γουρλωμάτις. Αυτό σημαίνει ότι το βασιλάκι διαγράφεται από αυτό τον κατάλογο. Βασιλάκι Boarfish. Ε, και η αιτιολόγηση είναι να λειτουργεί η απαγόρευση των απορρίψεων. Όχι, γίνεται δεκτή η προφορική τροπολογία. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 119. Τι συμβαίνει κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. η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 απορρίπτεται πέμπτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έκτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έβδομο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όγδο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ένα το τμήμα υπέρ να ελέγξουμε το 8ο τμήμα της 119 έναρξη του ελέγχου λήξη απορρίπτεται ένα το τμήμα της 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δέκατο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 240 υπέρ κατά αποχές έλεγχος της 240 έναρξη του ελέγχου λήξη απορρίπτεται τροπολογίες 293 και 301 με ονομαστική κλίση έναρξη λήξη συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Τροπολογία 264. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 227 με ονομαστική κλίση έναρξη λήξη εγκρίνεται 228 με ονομαστική κλίση έναρξη λήξη απορρίπτεται 216 με ονομαστική κλίση έναρξη λήξη απορρίπτεται τροπολογία 134 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 135 υπέρ κατά καταπίπτει, καταπίπτει κύριε συνάδελφοι περνάμε στην 135 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και καταπίπτει η τροπολογία 218 τροπολογία 265 υπέρ κατά αποχές θα την ελέγξουμε 265 έλεγχος έναρξη λήξη απορρίπτεται 241 με ονομαστική κλίση έναρξη λήξη εγκρίνεται Τροπολογία 139. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 266. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε τη 266, ε, έναρξη. Λήξη. απορρίπτεται τροπολογία 224 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία να ελέγξουμε τη 224 έναρξη του ελέγχου λήξη εγκρίνεται 267. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 157. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 285 με ονομαστική κλίση έναρξη. Λήξη. εγκρίνεται. Η τροπολογία 286 έχει αποσυρθεί. Περνάμε στην τροπολογία 230. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα το ελέγξουμε. 230 έλεγχος. Έναρξη. Λήξη. εγκρίνεται 242 με ονομαστική κλίση υπέρ κατά αποχές α, συγγνώμη, είναι ονομαστική κλίση λήξη εγκρίνεται 183 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 268 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 269 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 180 έλεγχος της 269 έναξη λήξη απορρίπτεται. Τροπολογία 185. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 287 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 270 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 225 με ονομαστική κλίση έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 226. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 243 με ονομαστική κλίση έναρξη. Λήξη. εγκρίνεται 197 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 288 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 302 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε στην ε, τροπολογία 298 με ονομαστική κλίση. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 202. Ποιοι είναι υπέρ. Ναι, κύριε Ρογκούτ. Παρακαλώ να επαναλάβετε την προηγούμενη ψηφοφορία. Ήταν ε, λάθος, ε, λάθος ο αριθμός στη μετάφραση. Την προηγούμενη ψηφοφορία να την επαναλάβετε παρακαλώ. Δεν μεταφράστηκε ίσως σωστά. You mean amendment 200... Εννοείται τη 271. Εντάξει. Ωραία. Ε, θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία για την τροπολογία 298. Ποιοι είναι υπέρ. So what was it? So we do 298 again. Ωραία. Επαναλαμβάνουμε την ε, ψηφοφορία επί της τροπολογίας 298 με ονομαστική κλίση. Έναρξη παρακαλώ. Λήξη. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 202. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 273. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε τη 273. Έναρξη του ελέγχου. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 219 με ονομαστική κλίση. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 231 με ονομαστική κλίση. Έναρξη. Λήξη. απορρίπτεται τροπολογία 232 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 223 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 233 με ονομαστική κλίση έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 274 ονομαστική κλίση έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 212 με ονομαστική κλίση έναρξη λήξη απορρίπτεται τροπολογία 289 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 213 καταπίπτει και περνάμε στην τροπολογία 276 με ονομαστική κλίση. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 234 με ονομαστική κλίση. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 244 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 277 έχει αποσυρθεί. Περνάμε στην τροπολογία 214 με ονομαστική κλίση έναρξη. Λήξη. απορρίπτεται τροπολογία 52 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 245 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε τη 245 έλεγχος επί της 245 έναρξη Λήξη. Εγκρίνεται. Θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο της πρότασης όπως τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέτω σε ψηφοφορία το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Έναρξη. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στην κυρία Ρώτης. Περνάμε στην έκθεση Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Ούσκη και εξετάζουμε την πρόταση κανονισμού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θέτω σε ψηφοφορία 53 τροπολογίες της... Η κυρία Ροτ Μπέρετ έχει ζητήσει το λόγο. Λοιπόν, 53 τροπολογίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Τις θέτω σε ψηφοφορία όλες μαζί. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος στη 48. Έναρξη του ελέγχου. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52 μονομαστική κλίση. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ελέγχουμε την τροπολογία 68. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Θέτω σε ψηφοφορία το αντίστοιχο τμήμα της τροπολογίας 49. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε Τροπολογία 49. Έναρξη του ελέγχου. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 51 κατά τμήματα με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα. Έναρξη. Λήξη. Παρακαλώ, ο εισηγητής έχει ζητήσει το λόγο. Ναι, κύριε Ουσκη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πριν την ψηφοφορία θα ήθελα να πω ως εισηγητής ότι αυτός, ο, αυτή η χωριστή ψηφοφορία δεν έχει έννοια εάν θέλουμε να αποφύγουμε ε, το μπέρδεμα ε, θα ήθελα να να ρωτήσω ε, εάν είναι δυνατόν αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν κατά του ενός τμήματος να καταψηφίσουν και τα δύο τμήματα. Ευχαριστώ. Uh, λοιπόν, συνεχίζουμε την ψηφοφορία ε, ε, όπως ακριβώς το έχουμε προγραμματίσει κατά τμήματα με ονομαστική κλίση. Ε, τροπολογία 51 λοιπόν, το πρώτο τμήμα, ψηφίσαμε και έχει απορριφθεί. Περνάμε στο δεύτερο τμήμα. Έναρξη. Let's repeat the vote on the first part of 15. Why? Uh, because there was some lack of clarity on the... Oh no, we're voting. Λήξη. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται και τα δύο τμήματα. Περνάμε στην τροπολογία 61 με ονομαστική κλίση. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Οι υπόλοιπε τροπολογίες καταπίπτουν και θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο της πρότασης όπως τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται θα θέσουμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σε ψηφοφορία το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική κλίση έναρξη λήξη Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Ούσκι. Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Τόρβαλτς. Και θέτω την έκθεση σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή θέτω σε ψηφοφορία το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική κλίση έναρξη Θα επαναλάβω λοιπόν την ψηφοφορία. Dear colleagues, I'm Ζητώ συγγνώμη αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον ρυθμό της ε, διερμηνίας. Ε, μπορείτε να δείξετε κατανόηση αν είναι δυνατόν. Για την έκθεση του κυρίου Τόρβαλτς, ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και περνάμε στην έγκριση του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Τόρβαλς. Περνάμε στην επόμενη έκθεση του κύριου Τόρβαλτς και την θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο της έκθεσης. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική κλίση, έναρξη, λήξη. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Τόλβαρτ και πάλι. Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Γκάλαχερ ο εισηγητής, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που στήριξε τον Εύρο και τον ε, ε, Ιανουάριο την, αναβολιά της, την αναβολή της έκθεσης για ε, γιατί ακριβώς θέλαμε να υπερβούμε το αδιέξοδο σε ό,τι αφορά τα μακροπρόθεσμα διαχειριστικά σχέδια μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Βέβαια, για αυτά τα διαχειριστικά σχέδια δεν έγινε πρόοδο μετά την εισαγωγή τη Σύνδεξη Λισαβόνα από το 2009 ούτε στη διάρκεια των διαδοχικών προεδριών. Ήταν όμως ακρογωνιαίος λήθος της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Στόχος των διαχειριστικών σχεδίων είναι να προστατεύσουν τους αλληλευτικούς πόρους και να εξασφαλίσουν και τη βιωσιμότητα ε, και την επιβίωση των κλάδων. Την προηγούμενη εβδομάδα επί Ιρλανδικής Προεδρίας το συζήτησαν οι Υπουργοί και ο Ιρλανδός Υπουργός επιβεβαίωσε στον πρόεδρό μας στον πρόεδρο της Επιτροπής δηλαδή Αλίας, Γκαμπριέλ Μάτο, ότι θα γίνει κάθε προσπάθεια ώστε να εξευρεθεί ένας αποδεκτός συμβιβασμός. Ως ένδειξη λοιπόν καλής έλυσης, η Επιτροπή Αλίας θα ήθελε πλέον να τεθεί σε ψηφοφορία σήμερα. Ωστόσο, προειδοποίηση σας απευθύνουμε, θα παρακολουθούμε και τις εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες. Και αν δεν σημειωθεί καμία πρόοδος, θα επανεξετάσουμε τη θέση μας και ίσως χρειαστεί να μπλοκάρουμε ε, ελπίζουμε να μην καταστεί απαραίτητο να μπλοκάρουμε ε, τι εξελίξει. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Υπάρχει διαδικαστικό από τον κύριο Λάγκεν. Παρακαλώ. Κυρία Αντιπρόεδρε, θα μπορούσατε να κλείσετε το τηλέφωνό σας ή να δώσετε τη θέση σας σε έναν σωστό πρόεδρο. Συνεχίζω με την ε, ψηφοφορία. Τα σχόλια εκφράζουν αυτούς που τα διατυπώνουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συνεχίζω με την ψηφοφορία. Λοιπόν, ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Γκάλαχε. Θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 34. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο της πρότασης της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εξετάζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο του νομοθετικού ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της πρότασης ψηφίσματος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 φράσεις οι οποίες ε, στην ουσία ε, δικαιολογούν την βία, κυρίως δέκατα των γυναικών. Μισογυνικές λοιπόν ε, συζητήσεις τις οποίες δεν μπορούμε να ανεχτούμε και ούτε ακόμα να τις δεχτούμε και επομένως μετεπιτάσεως ε, τις ε, καταδικάζουμε γιατί ε, δείχνουν και ένα είδος νοοτροπίας την οποία δεν μπορούμε να δεχτούμε εδώ γιατί διαφορετικά όλες οι συζητήσεις που κάνουμε εδώ πέρα θα είναι μάταιες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρησή σας. Περνάμε στην ψηφοφορία επί της πρότασης ψηφίσματος της Επιτροπής Γυναικών και Ισότητας των Φύλων σχετικά με την 57η Σύνοδο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη θέση της γυναίκας, εξάλληψη και πρόληψη κάθε μορφής βίας σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. Θέτω σε ψηφοφορία την παράγραφο 1 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4 κατά τμήματα με ονομαστική κλίση. Ναι. Πρώτο τμήμα, πρώτο τμήμα χωρίς ονομαστική κλίση. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα με ονομαστική κλίση. Έναρξη. εγκρίνεται. Παράγραφος 7 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση, έναρξη, λήξη, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 9, ποιοι είναι υπέρ, κατά,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 αιτιολογική σκέψη σίγμα τάφ κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο της πρότασης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε στην έκθεση, της κυρίας Λιωτάρ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη καινοτομία για την ενεργό και υγιή γύρανση. Θα την θέσω σε ψηφοφορία. Δεν έχουν υποβληθεί τροπολογίες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην πρόταση ψηφίσματος έξι πολιτικών ομάδων σχετικά με την 16η συνάντηση της διάσκεψης των συμβαλωμένων μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλληψη Άγριων Ιδών, Πανίδας και Χλωρίδας. Θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο της πρότασης. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση της κυρίας Χολμάιερ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2014. Θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 26 με ονομαστική κλίση, έναρξη. Λήξη. απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 με ονομαστική κλίση έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ποιοι είναι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω ότι η συγγήτρια έχει ζητήσει το λόγο για να προτείνει μια προφορική τροπολογία η κυρία Χολμάιερ Κυρία ε, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η προφορική τροπολογία θα είναι σύντομη. Το demand driven υποκαθίσταται από το end και το ε, επόμενο κείμενο παραμένει ως έχει. Επίσης, επί της προφορικής τροπολογίας της κυρίας Χολμάιερ γίνεται δεκτή, οπότε θέτω σε ψηφοφορία την παράγραφο 6 υπέρ. Είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση έναρξη λήξη απορρίπτεται τροπολογία 15 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την τροπολογία 24 έναρξη του ελέγχου παρακαλώ λήξη εγκρίνεται τροπολογία 17 με ονομαστική κλίση έναρξη λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογίες 20 και 27 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος με ονομαστική κλίση έναρξη λήξη εγκρίνεται και περνάμε στην έκθεση του κυρίου Μπαλντασάρε σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη Θέτω σε ψηφοφορία την παράγραφο 5 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 17 κατά τμήματα και με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 26 κατά τμήματα με ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, έναρξη. λήξη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 30. Πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 42. Μονομαστική κλίση. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 47 Πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ο εισηγητής, ο κ. Βαλτασάρε, έχει ζητήσει το λόγο για να παρουσιάσει μια προφορική τροπολογία. Μετά την παράγραφο 47 θα πρέπει να γραφτεί το εξή Θέματα συμμόρφωσης και σχέσει με τι τρίτες χώρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει αντίρρηση. Περνάμε λοιπόν στην ε, ψηφοφορία τη παραγράφου. Ωραία. ψηφίζουμε την ε, ε, πρόταση που παρουσίασε ο εισηγητής ο κύριος Μπαλτασάρε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Παλτασάρε. Και περνάμε στην έκθεση του κυρίου Χάουιτ σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Θέτω σε ψηφοφορία την παράγραφο 3 με ονομαστική κλίση έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Μονομαστική κλίση έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 13. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 21 υπέρ okay. we'll check paragraph 17 ελέγξουμε την παράγραφο 17 λήξη απορρίπτεται παράγραφος 21 είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 26 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 29 με ονομαστική κλίση έναρξη λήξη εγκρίνεται παράγραφος 31 με ονομαστική κλίση έναρξη Α, ναι. Ε, λήξη εγκρίνεται. Παράγραφος 33 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 36 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 38 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 40 ονομαστική κλίση έναρξη λήξη εγκρίνεται παράγραφος 44 ονομαστική κλίση έναρξη Λήξη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 45. Ονομαστική κλίση έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 56. Υπέρ να ελέγξουμε την παράγραφο 53. Έναρξη του ελέγχου. Λήξη. Απορρίπτεται. Παράγραφος 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 67 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 73 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος στο δεύτερο τμήμα της παραγράφου 73 έναρξη λήξη απορρίπτεται παράγραφος 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 84 μονομαστική κλίση έναρξη λήξη εγκρίνεται παράγραφος 85 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 86 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 87 παράγραφος 86 δεύτερο τμήμα έλεγχος έναρξη λήξη εγκρίνεται. Παράγραφος 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 91 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Β υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη σίγμα τάφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, νομίζω ότι είναι καθαρό το αποτέλεσμα αιτιολογική σκέψη J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη Ι, δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και θέτω σε ψηφοφορία το σύνολο της πρότασης ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Χάουιτ is the, the explanation